του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και από την ομάδα των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων έχω κάποια αιτήματα για ορισμούς επιτροπών και κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών και ο κατάλογος των διορισμών θα, μπουν, θα μπει στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση στα πρακτικά θα θεωρήσουμε ότι έχουν επιβεβαιωθεί αυτοί οι διορισμοί. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος μα έχει